If Καθίστε παρακαλώ, για να μπορέσουμε και να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο σημείο της ημερίας αδιάτραξης, που είναι ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της ΕΑΤ, Θέλουμε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία γιατί έχουμε διαφορετικό αριθμό μελών αυτή τη στιγμή απέναντί μας. Είστε μόνο τα μέλη της ε, ΕΚΟΝ. Λοιπόν, ξεκινάει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Λοιπόν, κάποια μέλη καθυστέρησαν Δύο ε, περισσεύουν από το ΕΛΚ. Ένας τώρα περισσεύει από το ΕΛΚ. Ωραία. Ακόμα πέντε συνάδελφοι δεν έχουν έρθει. Ωραία, λοιπόν, τελείωσε η δοκιμαστική ψηφοφορία. Μπορούμε λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε για το διορισμό του Τζέρι Κρός ως εκτελεστικό διευθυντή της ΕΑΤΣ για μια πενταετή θητεία είναι ε, μυστική ψηφοφορία, ε, ξεκινά. Πέρας. 24 υπέρ, 27 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. Machado. No, I need to, I need to know exactly the name of the person we are voting. Okay. Are we sure? Yes. Okay. Now we move on to the next vote. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία που είναι ο διορισμός του Πέδρο Ματσάδο ως μέλους του ενίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για πενταετή θητεία και πάλι μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας δεν έχει ψηφίσει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται αυτός ο διορισμός. Περνάμε τώρα στον επόμενο διορισμό του κυρίου Σουρίνα, Ω μέλου του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης για πέντε χρόνια, μυστική ψηφοφορία και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «43 υπέρ, 5 κατά, 4 αποχές, εγκρίνεται». Περνάμε τώρα στο διορισμό του Ζαν Καρπεντιέ ως αντιπροέδρο του ενιαίου Συμβουλίου Εξηγένση για πενταετή θητεία και πάλι είναι μυστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 37 υπέρ, 11 κατά, 5 αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων για τον κανονισμό και την, ε, για την εξηγίαση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας. 48 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Okay. Sorry, but now we... Ωραία, λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ετήσια έκθεση για το 2018. Εισηγητή ο κύριος Μαυρίδη. Ξεκινάμε, λοιπόν, με το αρχικό κείμενο ε, υπό ένα ε, άρχεται ψηφοφορία. Oh, I'm sorry. I was just... Με συγχωρείτε, εγώ βιάστηκα, ε, συγχωρέστε με. Against. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Uh, compromise. Συμβιβαστική α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στη συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας πέρας 22 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Ένα έλκε παραπάνω. Σωστά. Ακόμα περισσεύει ένα, μια ψήφιση από PPP. Από το ΕΛΚ, συγγνώμη. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Mm, απορρίπτεται. 26 υπέρ, 27 κατά. 130 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται subheading 2 ε, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ήττα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 175 έναρξη ψηφοφορίας. Ένα ΕΛΚ περισσεύει. Πέρας. 17 υπέρ, 32 κατά, 4 αποχές απορρίπτεται. 177 ε, υπέρ, κατά, αποχές, να ξαναελέγξουμε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22, 30, απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 208 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 συγγνώμη 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Συμβιβαστική ελέη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική λάμδα υπέρ μη συγγνώμη αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 242 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβεβαστική Q υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική R. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται. Συμβιβαστική It was approved, Louis. Είχε εγκριθεί, Λουίς. Συμβιβαστική S. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΣΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 277 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπάρχει μια προφορική τροπολογία από τους πράσινους. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις... Ναι, Μάρκους. Ε, αφού ψηφίσαμε ε, το προηγούμενο, μου φαίνεται λίγο δύσκολο εδώ. Γι' αυτό το λόγο εμείς ως ΕΛΚ ε, δεν θα το ψηφίσουμε αυτό. Είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας. Not to put it to the vote. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί. So how many people are against? Πώς είναι κατά. Ποιοι είναι κατά του να ψηφιστεί. Είναι πάνω από τέσσερις, οπότε προχωράμε. So, we move on to amendment 200. Πάμε στη 299 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην παράγραφο 22, το αρχικό κείμενο του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη ε, συμβιβαστική Y, στις ιδεολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z, Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη ε του εισηγητή αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 κατά αποχές απορρίπτεται. 45 44, συγγνώμη, 45, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε στο αρχικό κείμενο στο σημείο αναφορά ένα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική χ υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Σημείο αναφορά 4. Ε, αρχικό κείμενο του εισηγητή υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογική αναφορά 6 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 7 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ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 Okay. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Εκεί θα ψηφίσουμε για την απαλλαγή του 2018 για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Παράγραφος 1, τροπολογία 1, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Έχουμε και μία προφορική τροπολογία εδώ. Έπινγκ. Έχουμε αντιρρήσει. Μπορούμε να ψηφίσουμε και την προφορική τροπολογία επινκ. Ωραία. Υπέρ αυτή. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Εδώ θα ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Με συγχωρείτε, διορθώνω. Περνάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά άποχες Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλω να το δούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ στην 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Με συγχωρείτε. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 15. Θα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 16. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε το μέσο. στην τροπολογία υπερθμών 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο όπως τροποποιήθηκε, ονομαστικά παρακαλώ, Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στην απαλλαγή τη ΕΙΟΠΑ, τη Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Παράγραφος 1. Υπέρ, κατά, α, τροπολογία 1 διορθώνει η πρόεδρο. Τροπολογία αριθμό 1, στην παράγραφο 1. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την ε, τροπολογία αριθμός 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 28 υπέρ, 23 κατά. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Εγκρίθηκε. 28 υπέρ, 17 κατά και 5 αποχές. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εδώ πρέπει να ελέγξουμε. Τροπολογία 15. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. 22 υπέρ, 26 κατά. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο συνεπώς. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Ψηφίζουμε τώρα το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 48 υπέρ, 3 κατά. Εγκρίθηκε. Τώρα, συνεχίζουμε και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία που είναι η απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ΕΣΜΑ. Τροπολογία αριθμός 1, παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Α, όχι, 6, 6 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εδώ πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ.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 23 ναι, έχει και δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 48 υπέρ, 2 κατά. Εγκρίθηκε. One minute and then we move to the next. Ωραία, συνεχίζουμε τότε και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι πολιτική ανταγωνισμού ετήσια έκθεση. Σε ένα λεπτό παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. So thank you. We have now point... Είμαστε στο σημείο 23, πολιτική ανταγωνισμού τώρα. Ετήσια έκθεση 2019. Η συγκεκριά μας είναι η Στεφανή Ιον Κουρτά. Της δίνω και το λόγο λοιπόν για πέντε λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ Στεφανή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ναι, καλημέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, που βοήθησαν για τη συνεργασία τους και για την συνεισφορά τους στην έκθεση αυτή. Έχουμε 345 τροπολογίες που υποβλήθηκαν και πολύ χαίρομαι που θα μπορέσω να συνεργαστώ μαζί τους για να καταλήξουμε σε τροπολογίες συμβιβαστικέ. Η κυρία Βεστάγκερ, η Επίτροπος, είπε ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί προτεραιότητα της τωρινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε πολύ χαίρομαι για αυτό το φιλόδοξο χάρτη πορείας. Και χαιρετίζω εδώ και την παρουσία του νέου Γενικού Διευθυντή ε, για τον ανταγωνισμό, που το γνωρίζουμε βέβαια από παλιότερα, τον Ολιβιέ Γκαρσό. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Μπορούμε λοιπόν, πιστεύω, να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των διάφορων πολιτικών ομάδων μας εδώ για το ότι θέλουμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού και ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να λάβουμε υπόψη μας τους στόχους της ε, Πράσινης Συμφωνίας, τον ηλικιώδη ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται η ψηφιακή τεχνολογία και επίσης την ε, ακαιρεότητα της αγοράς. Ευχαριστώ την Άγκρε, την Ίντα, την Ίμκο για τις νομοδοτήσεις τους που θα λάβω υπόψη μου στην εκθεσή μου. Ε, θα επανέλθω λίγο στα κύρια σημεία που τονίζω με τους κοιόδης εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και θα ξεκινήσω από το ΕΛΚ. Ναι, συμφωνώ με τη βούληση του ΕΛΚ να έχουμε μεγαλύτερη αμοιβαιότητα με τρίτες χώρες ώστε να διασφαλίσουμε αυτή τη, αυτές τις ισότιμες συνθήκες για τις επιχειρήσεις μας. Ε, στα ψηφιακά συμφωνώ ότι πρέπει να σταματήσει το self-preferencing που έχουν ορισμένες πλατφόρμες και συμφωνώ επίσης και με την βούληση να ξαναδούμε λίγο το δόγμα της διευκόλυνσης με τα ψηφιακά, όπως επίσης και την ανακοίνωση για το ΡΟΜΕΤ που νομίζω ότι χρειάζεται ανανέωση, δεδομένου ότι οι ψηφιακές αγορές εξελίσσονται ταχύτατα. Επίσης, θέλω να προσφέρω περισσότερη νομική ασφάλεια στι επιχειρήσει, όπως και εσείς υπογραμμίζετε, προκειμένου να έχουμε ένα σχέδιο συνεργασίας για να ενισχύσουμε την συμμετοχή και την ε, εμπιστοσύνη. Ε, στρέφουμε στους σοσιαλιστές. Αγαπητή Κάρμεν, ε, βλέπω ότι πάνω από 15 τροπολογίες συνυπογράφουν το ΕΛΚΑ και οι σοσιαλιστές. Κάτι δείχνει αυτό. Και εμείς συμφωνούμε ότι όντως υπάρχει η ίδια διάγνωση από όλες τις πλευρές όσον αφορά τα ψηφιακά και τον ανταγωνισμό. Κυρίως για αυτά που λέτε για τα δεδομένα, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την οικονομία των δεδομένων, να δούμε τη διαλειτουργικότητα για το πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να ξαναδούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού, για να εξετάσουμε ε, το σημαντικό αυτό φαινόμενο της συγκέντρωσης, της συσσόρευσης και της χρήσης των δεδομένων όταν γίνονται συγχωνεύσεις. Έπειτα, η αξιολόγηση εξάντε πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τα διάφορα μοντέλα που λειτουργούν στην ψηφιακή οικονομία, ώστε γίνεται πιο γρήγορα να εντοπίσουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού και να μπορέσουμε να δράσουμε έγκαιρα από την αρχή όσο προλαβαίνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσφύγουμε σε αυτά τα εξάντε μέτρα στην ψηφιακή αγορά, γιατί όσε επιχειρήσει έχουν δεσπόζουσα θέση είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Επίση, χαιρετίζω και την τροπολογία που ζητάει η Γενική Διεύθυνση Κόμου να έχει εμπειρογνώμονε στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι να επανδρώσουν τι ε, ήδη υπάρχουσε ε, ομάδε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα και να αξιολογήσουμε πλήρως τα ζητήματα συνδεσιμότητας που τίθενται ε, μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων που δεσπόζουν την αγορά. Επίσης, θέλω να έχουμε πιο συχνά ανταλλαγή απόψεων με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κυρίως μέσω της ομάδας εργασίας ανταγωνισμού της δικιάς μας Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. Στρέφομαι στους πράσινους τώρα. Σβέν, αγαπητέ Σβέν, όπως ε, και όλοι ευχόμαστε να πετύχει η πράσινη συμφωνία της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Και σημείωσα τις τροπολογίες των πρασίνων, που δεν είναι οι μόνες, αλλά υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να λάβουμε υπόψη μας τους στόχους της πράσινης συμφωνίας στην επόμενη αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές επιχορηγήσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες αυτές με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάργηση του άνθρακα και προστασία του κλίματος. Επίσης, όπως και άλλοι πιστεύω και εγώ, ότι πρέπει να δούμε τα κατόφλια των ε, αποκτήσεων ε, επιχειρήσεων για να ξέρουμε ποια είναι τελικά η αξία της συναλλαγής στο σύνολό της. Στρέφομαι στην ΚΟΕ τώρα. Γενικά μιλώντας, δεν ξέρω αν είναι εδώ και ο δισηγητή. Όπω είπα και νωρίτερα, η πολιτική ανταγωνισμού πιστεύω ότι έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για την επιτυχία τη Πράσινη Συμφωνία, αλλά και στην παγκοσμιοποίηση για να πετύχουμε αυτή την ισότιμη αντιμετώπιση αλλά συγχρόνω πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε την ακερότητα τη αγορά μα. Όλοι μας θέλουμε πολιτική για την πολιτική ανταγωνισμού, προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική, να εφαρμόζει σωστά τους κανόνες και μπορεί όντω να κάνει πολλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τα πάντα. Τώρα, να μιλήσω λίγο για τις τροπολογίες όσον αφορά τη φορολογία. Η Γκουε ε, κατέθεσε τέτοιες τροπολογίες. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν συνδέεται άμεσα με τη φορολογική πολιτική, γιατί οι κανόνε ανταγωνισμού δεν μπορούν να παρέμβουν στη βαρολογική πολιτική που είναι εθνική. Παρ' όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμέ να βοηθήσουμε τις χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει ότι πρέπει να υπάρχει ευνοϊκή αντιμετώπιση των επιχειρήσεων, αλλά συγχρόνω, πιστεύω και η Επίτροπος Βαστάγκερ έδειξε το θάρρος της και την επιμελιά της επ' αυτού να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση της Apple. Επίσης, γνωρίζω ότι και η Επίτροπος αλλά και εσείς θέλετε να τη φόροι εκεί που δημιουργούνται τα κέρδη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφαθεί από αυτού και έχει ψηφίσει την έκθεση σε ΣΕΤΕΜΠΕ. Τέλος, αγαπητή Φρανσίσκα, ευχαριστώ την ομάδα σας που θέτει την προβληματική των ισιωτικών περιοχών. Είναι αλήθεια ότι το χαρακτηριστικό αυτό του νησιού μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες και μπορεί να οδηγήσει σε εμπόδια στον ε, θεμητό ανταγωνισμό στην εθνική αλλά και στη διεθνή αγορά. Τα νησιά, και ξέρουμε ότι έχουμε πολλά νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ένα μειονέκτημα ανταγωνιστικό και για την προμήθεια ενέργειας και για τις μεταφορές, αλλά και για τις υπηρεσίες ακόμα που είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα σωστά. Να λοιπόν κάποια πρώτα στοιχεία μετά τις ανταλλαγές που είχα με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε την ανταλλαγή αυτή και γι' αυτό περιμένω πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις από σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Στεφανή για την εισαγωγή που έκανες. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις. Έχουν τέσσερα λεπτά ο καθένας από το ΕΛΚ, ο Στέφαν Μπέρκ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο, πιστεύω ότι και εγώ 335 τροπολογίες δείχνουν ότι η εκθεσή αυτή αποτελεί τη βάση για τα όσα θα κάνει η Κομισιόν μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αυτός, αυτό το πλήθος ε, τροπολογιών υπογραμμίζει πόσο σημαντική αυτή είναι η έκθεση για τον ανταγωνισμό σε αυτή την ε, περίοδο. Πιστεύω επίσης ότι είναι καλό ότι πολλές ενδιαφέρουσε τροπολογίες ε, ε, παρατηρούμε. Αυτές δείχνουν την κατανόηση, την αναγνώριση του ότι έχει αλλάξει ο κόσμος και ότι και στην πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες, ε, τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα για τις νέες δομές, ε, τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Ο εισηγητής ήδη ανέφερε κάποια σημαντικά θέματα. Πρώτον, βρισκόμαστε σε μια φάση που πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο τα κατόφλια που έχουμε είναι ακόμα σε ισχύ. Είναι συναρπαστική η συζήτηση ε, αυτή που θα κάνουμε στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε τις ψηφιακές αγορές, ε, ε, gatekeeper, αλλαγμένες δομές αγοράς, νέες δομές αγοράς και εκεί πρέπει να αναρωθούμε για τα δεδομένα, για τις τράπεζες δεδομένων. Θα πρέπει να αποτελεστώ αντικείμενο εντατικότερης διαπραγμάτευσης. Επίσης, το name and shame ως αρχή πρέπει να το δούμε ξανά από διάφορες απόψεις Γενικότερα, θεωρώ ότι αν ε, ε, βλέπουμε τα πράγματα εκ των προταϊρών, ε, κάποια πράγματα θεωρείται ότι έχουν νόημα, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολικά πολλά. Να μην στείλουμε λάθος σήματα στις εκάστοτε επιχειρήσεις. Να βλέπουμε δηλαδή κατά πόσο πρέπει να δραστηριοποιείται αμέσως η Κομισιόν ή πρώτα να βλέπει την οικονομική κατάσταση και μετά ε, να βλέπει, να εκδίδει εκθέσεις. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες που θα αποσχολήσουν εμά τις συζητήσει μας. Πιστεύω ότι κατά βάση η έκθεση είναι εντάξει. Μπορεί να δώσει απαντήσεις στις νέες ερωτήσεις και στα προβλήματα και αναμένω τις ε, επερχόμενες διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Berger, for... Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέργκερ. Η Κάρμεν Γκαμπριέλα Αραμέχη το λόγο από τους σοσιαλιστές. Αγαπητή Στεφανή, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσα εμπειρία. Είναι η πρώτη μου έκθεση για την ΕΚΟΝ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την εξαιρετική συνεργασία μέχρι τώρα. Όπως είπα όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο έκθεσης είναι καλή και προσπαθώ απλώς να την βελτιώσω σε κάποια σημεία τα οποία θεωρώ πως αυτό θα χρησιμεύε και χαίρομαι που πολλές από τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα τις συμπεριλάβατε. Όπως είπε και η Στέφανη, θα ήθελα να μιλήσω για τις τροπολογίες, για τη συγκέντρωση και χρήση και συλλογή των δεδομένων σε περίπτωση ε, διατάξεων antitrust, όπως επίσης όπου ισχύει η νομοθεσία περί συγχωνεύσεων. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε για να καταλάβουμε την ενδεχόμενη ή δυνητική ε, αρνητική επίδραση που θα έχουν στις νέες επιχειρήσεις που προσπαθούν να μπουν και να γίνουν ανταγωνιστικές σε συγκεκριμένη αγορά. Εδώ προσπάθησα να ενισχύσω την ιδέα πως δεν υπάρχουν ε, δωρεάν υπηρεσίες. Εμείς με τα προσωπικά μας δεδομένα πληρώνουμε πολύ ακριβές υπηρεσίες. Γιατί τα δικά μας δεδομένα έχουν γίνει το πετρέλαιο του σήμερα, όπως λένε κάποιοι. Οπότε οι ρυθμιστέ, οι νομοθετέ κατάλαβαν πως τα πρόστιμα δεν λύνουν την περίπτωση. Είναι απλώς ένα κομμάτι του κόστους που απορροφούν ε, στα πλαίσια του συνηθισμένου επιχειρήν οι γίγαντες της τεχνολογίας. Και η αναγνώριση προσώπου, όπω επίση και η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν ξέρω αν εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια προφορική τροπολογία αργότερα και να αναφέρουμε την συλλογή δεδομένων μέσω τεχνικών αναγνώρισης προσώπου και των κινδύνων που ελοχεύουν. Επίσης η τροπολογία που αναφέρεται στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πλήρως ε, πρικοδοτημένη με εμπειρογνώμονε σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να καταλάβουν καλύτερα ποια είναι τα διορθωτικά μέτρα τα οποία θα είναι όλο και πιο επιτακτικά να λάβουμε στο μέλλον. Επίσης, τροπολογίες για τον κλάδο offline, δηλαδή σούπερ μάρκετ, διανομή, και για τις ρουμανικές τράπεζες, 2,95 είναι η τροπολογία, η κίνδυνη της συμπεριφοράς και της δημιουργίας καρτέλ. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία και στα κλειστά οικοσυστήματα, για παράδειγμα αυτό της Apple, και να μιλήσω και για την αναθεώρηση του ορισμού της αγοράς που όλοι καλωσορίζουμε τέλος να μιλήσω για την τροπολογία 3.10, την οποία όλοι καλωσορίζουμε. Θέλουμε περισσότερη ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών πέραν του δομημένου διαλόγου με την κυρία Μπεστάγκερ στο Κοινοβούλιο, γιατί ε, εκπροσωπούμε 550 εκατομμύρια ε, καταναλωτές. Χρειάζεται λοιπόν στην ομάδα εργασίας ανταγωνισμού στην ΕΚΟΝ να κάνουμε περισσότερες ανταλλαγές ε, απόψεων και με την κυρία Επίτροπο και με τη Γενική Διεύθυνση. Θα ήθελα να συνεργαστούμε για αυτό το τόσο ενδιαφέροντα φάκελο. Προσδοκώ πως θα είναι καλή η συνεργασία και πως με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε και τους καταναλωτές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ο Σβέν Κίκολτ ε, για, τον, για τους πρασίνους, όπου δεν είναι σίγουρα η πρώτη του έκθεση εδώ. Τέσσερα λεπτά για σένα Σβέν και παρακαλώ να αναλάβει για μερικά λεπτά η Στεφανή την Προεδρία. Λίγες παρατηρήσεις από πλευράς μου. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που βλέπετε θετικά τις τροπολογίες μας ε, για να συμπεριληφθεί η Πράσινη Συμφωνία στην έκθεση. Αναμένουμε με ανυπομονησία για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, διότι θεωρούμε ότι θα έχει σημαντικέ συνέπειε για την πολιτική ανταγωνισμού η έγκριση αυτών των τροπολογιών. Αυτό συνάδει και με την ανακοίνωση τη Κομισιόν ότι όλοι οι κανόνε και οι κανονισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν συνοχή με του στόχου τη πράσινη Συμφωνία. Οπότε α τι εξετάσουμε επικοδομητικά. Δεύτερον, παρατηρώ στην εξάντε monitoring, την εξάντε παρακολούθηση και το σχετικό ζήτημα και όσον αφορά τις πλατφόρμες και όσους έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά βλέπω διάφορες αντιφατικές τροπολογίες και από τη δική σας οικογένεια Στέφαν Μπέργκερ οπότε αναμένω να δω ποια από τις διαφορετικές φωνές τελικά που ακούμε είναι η πραγματική ordnance πολιτική αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η παρακολούθηση εξάντε δεν είναι ε, ε, κατάχρηση κρατικής ε, εξουσίας όταν υπάρχει ολογοπόλιο ή μονοπόλιο και αν υπάρχει μονοπόλιο δεν καταλαβαίνω γιατί η παρακολούθηση εξάντε δεν συνάδει με την οικονομία, της κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αν υπάρχει μονοπόλιο λοιπόν υπάρχουν καλά επιχειρήματα που μας λένε ότι αν επιτρέψουμε να υπάρχει τέτοιο μονοπόλιο για λόγους ε, ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει σωστός ανταγωνισμός διότι θα ε, η μία μόνο πλατφόρμα δημιουργεί επαρκή δικτύωση, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία για όσους τη χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν ε, το, η εξάντε παρακολούθηση της αγοράς έχει νόημα και ήθελα επίσης να πω υπάρχουν και παρόμοιες ιδέες από την εισηγήτρια ότι ε, σε ψηφιακές εποχές η Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτεί να φτιάξει μια εποπτική αρχή. διότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια ψηφιακή κοινή ψηφιακή αγορά με 27 διαφορετικές δικαιοδοσίες με μικροδιαφορές ε, στην εφαρμογή της νομοθεσίας πλαισίου. Αυτό δεν θα βοηθήσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, δεν θα μας βοηθήσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού και ούτε θα μας βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή Ευρώπη βάσει των παραδόσεων της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Οπότε θα ήταν καλό το μήνυμα που θα δίναμε ε, δημιουργώντας έναν ενιαίο ψηφιακό επόπτη. Και τέλος ήθελα να πω και αυτό ίσως είναι το βασικό θέμα της έκθεσης, το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζουμε τις προφανείς διαφορές μεταξύ των δικών μας προτύπων και των προτύπων των τρίτων χωρών είναι σημαντικό. Χαίρομαι που η εισηγήτρια εστιάζει την προσοχή σε αυτό. Και φυσικά η υπόθεση Siemens Alstrom ήταν αυτή που πυροδότησε τη συζήτηση αυτή. θα μπορούσαμε καλύτερα να απορρίψουμε την αξία της σκληρή, του σκληρού ανταγωνισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γίνεται εδώ ακριβώς, λένε ε, εδώ κάποια κομμάτια του κειμένου ότι μπορείς να ανταγωνιστείς παγκοσμίω μόνο αν έχεις σκληρό ανταγωνισμό στη δική σου εσωτερική αγορά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί παγκοσμίω ε, εφαρμόζοντας σκληρό ανταγωνισμό εντός της κοινή αγοράς. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αυτό ως κοινό κανόνα. Απαιτείται ανάλυση σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κλάδο. Και σε ορισμένες περιπτώσεις Ορισμένοι από τους κανόνες μας ε, ε, δημιουργούν βλάβη στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά η γενική αρχή θα πρέπει να είναι ότι θέλουμε να έχουμε ισχυρό ανταγωνισμό ε, μεταξύ εταιριών υπό ένα κοινό κανόνα πλαίσιο. Σε κάποιες διατυπώσεις εδώ πέρα στο κείμενο το τραβάμε πολύ. Ε, ισχυριζόμαστε ότι ο ανταγωνισμός εντός της ευρωπαϊκής αγοράς μεταξύ ευρωπαϊκών εταιριών δημιουργεί πρόβλημα στη δική μας ανταγωνιστικότητα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια συμβεστική για να καταφέρουμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Okay, thank you, Sven Giegold. So, uh, Ευχαριστούμε, Sven Giegold. Uh, replace, um, Αντικαθιστώ τον πρόεδρο. Ε, τώρα όμως πρέπει να απαντήσω μια που πρόκειται για την έκθεσή μου. το συγγνώμη αν ε, δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα, αλλά μετά τέσσερα λεπτά η ε, επόμενη. Η κυρία Ντονάτο. Μάλλον δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Εκτός μικροφώνου της ομιλήτρια. Is it okay? Okay. Τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, έλεγα, είμαι ικανοποιημένη για το πνεύμα συνεργασίας και την συνεννόηση με τους συναδέλφους και τις κοινέ απόψεις όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης και τις τροπολογίες. Ειδικότερα, συμμερίζομαι την παρατήρηση που ακούσαμε πριν λίγο, ότι είναι σημαντικό να δώσουμε προσοχή στον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών εταιριών σε σχέση με τις χώρες εκτός Ευρώπης. Μερικές φορές φαίνεται οι κανόνες ε, του ανταγωνισμού εσωτερικά να υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των δικών μας εταιριών στην παγκοσμία αγορά, όπου καλούμαστε να ανταγωνιστούμε κολοσσούς. Και φυσικά τώρα μιλάμε για τους Κινέζους, κινέζικους κολοσσούς, αυτούς αναφερόμαστε, οι οποίοι δεν έχουν καμία τροχοπέδη όσον αφορά κρατικές επιχορηγήσεις πολύ υψηλές. Η ευκαιρία να θεωρήσουμε τώρα τους κανόνες για τις κρατικές επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να μην τιμωρούνται οι δικές μας ε, εταιρείε ε, στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, είναι πάρα πολύ σημαντική και κατεπίγουσα. Η εσωτερική ανταγωνιστικότητα, ο εσωτερικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κατά την άποψή μου να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την αρχή της ισότητας και της ισορροπίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Διότι είμαστε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δεν είμαστε απλή αγνή οικονομία της αγοράς όπου δεν λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πτυχή. λαμβάνεται υπόψη και η κοινωνική πτυχή και η απασχόληση. Ειδικότερα αναφέρομαι στο ότι είναι αναγκαίο να προστατεύουμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και των δημοσίων επιχειρήσεων στην αγορά και ότι πρέπει να προστατεύουμε τις startup ε, από το να τις καταπιούν οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Τέλος, ήθελα να επαναλάβω αυτά που έχω συμπεριλάβει στη δική μου τροπολογία, ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνετε υπόψη επίσης και το... Να λαμβάνετε υπόψη επίσης τα... οι ελλείψεις ανταγωνιστικότητας ορισμένων περιοχών σε σχέση με άλλες και αναφέρομαι ειδικότερα τώρα στις νησιωτικές περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν οι κρατικές ενισχύσεις ε, να παρέχονται όταν μιλάμε για επενδύσεις σε νησιωτικές περιοχές ή σε περιοχές γενικότερα μειονεκτούσες από άποψη δομική σε θέματα ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες, ούτως ώστε να έχουμε μια ανάπτυξη ομοιογενή ε, σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Κατά την απόψη μου επίσης, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε ούτως ή άλλως στις χώρες τη δυνατότητα golden share σε τομείς ε, σημαντικής ε, εθνικής κυριαρχίας ε, και στρατηγικής. Αλλιώς δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε τους βασικούς τομείς για κάθε χώρα σε αυτές τις βασικές πτυχές. Ελπίζω να έχουμε όλο και μεγαλύτερη σύγκληση απόψε. Ευχαριστώ. Sorry. Thank you, Francesca. Ραφαέλα Φίτο. Ή ή κάποιος άλλος από το ECR. Είναι εδώ κάποιος? Όχι. Μανού Αμπρί. Γκουε. Δεν είναι. Άρα όλοι συμφωνούν με την έκθεσή μου. Τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα. Catch the eye. Ερωτήσεις. Τρεις από το ΕΛΚ. Νίμκοτ Φιτζέραλτ και Ανδρέα Σουάπ. Παρακαλώ. Ένα λεπτό καθένας, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, λέει κυρία Γκιόρη. Ήμουνα ε, συγκήτρια από πλευρά στη ΣΥΝΤΑ, συντάκτρια γνωμοδότησης ουσιαστικά. Και έχω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερα για να πετύχουμε την ισότιμη μεταχείριση βασικανόνων στο πολυμερές ε, σύστημα εμπορίου. Και αυτή είναι η πτυχή που θέλησα να υπογραμμίσω με τις τροπολογίες που υπέβαλα, όπως επίσης και στην γνωμοδότηση της ΣΥΝΤΑ. Δεύτερον, βιομηχανική πολιτική. Δύο παρατηρήσεις έχω εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, ωραία. Δεν σημαίνει όμως χαλάρωση του ανταγωνισμού και ούτε να είναι σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν και το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού ΕΠ. Δεν θα πρέπει να πληγούν αυτές. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να δυσδύουν σε νέες αγορές με ένα φιλικό εμπορικό περιβάλλον. Και τέλος... για το λεγόμενο killer acquisitions, την απόκτηση δηλαδή με σκληρό τρόπο επιχειρήσεων και εκεί πρέπει να υπάρχουν κανόνες και να μην είναι τόσο εύκολο τις νοσίστατες επιχειρήσεις να τις παίρνουν οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις που δεσπόζουν στην αγορά γιατί έτσι εξαφανίζεται η δημιουργικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να τονιστεί και να φροντίσουμε τα προϊόντα των μικρομεσαίων να πολλούνται. Δεν πρέπει να αποτελεί κίνητρο αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Stephanie, thank you for your work uh, on this file, uh, which I think... Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστή η κατεύθυνση που ακολουθεί η έκθεση, αλλά ένα σημείο θα ήθελα να αναφέρω. Παράγραφος 13. Με εκπλήσει κάπως γιατί καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσει την ε, προσωρινή της έκθεση ε, για το Spotify και την καταγγελία εκεί και αν θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας πάνε στα σοβαρά, δεν θα πρέπει να προδικάσουμε εμείς μια έρευνα η οποία βασίζεται σε νομική καταγγελία κατά εταιρεία. Θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει με τη δέουσα επιμέλεια και να μην παρεμβαίνουμε ε, χωρίς λόγο. Βεβαίως η έρευνα θα πρέπει να τελειώσει το νωρίτερο δυνατόν, αλλά για να ζητήσουμε να κινηθεί η ε, διαδικασία, η νομική διαδικασία, όταν ακόμα δεν έχει καταλήξει η έρευνα, μου φαίνεται υπερβολικό. Θα ήθελα να με εξηγήσει η συγγήτρια τι πιστεύει και να το ξαναδεί. Ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά. Προφανώ στην έκθεση υπάρχει, έχουμε και πολύ καλό περιεχόμενο, αλλά νομίζω ότι κάποια ερωτηματικά ε, υπάρχουν και σα παρακαλώ σκεφτείτε τα και ε, απαντήστε μου για, τις, για τα ζητήματα που σα έθεσα. Ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας, ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια Στεφανή για τα όσα έχεις κάνει. Πιστεύω πως είναι εξαιρετική αρχή και είμαι πολύ περήφανος που ο Στέφαν Μπέργκερ ε, υπέβαλε τις τέλειες τροπολογίες, τις οποίες πλήρως ε, στηρίζω. Ένα θέλω να πω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Κάρμεν ε, Αβραμ που συνυπογράφει την τροπολογία με εμένα και το λέω για να το ακούσει και ο Γενικός Διευθυντής. Συζητάμε τις υποθέσεις επιχειρήσεων που δεν θέλω να κατονομάσω γιατί όπως είπε η συνάδελφος προηγουμένως δεν πρέπει να αναφερόμαστε ρητά σε επιχειρήσεις, αλλά εδώ η, η εταιρεία στην οποία αναφέρομαι έχει περάσει ήδη από τρεις έρευνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν πληρώσει ψηλά πρόστιμα. Ο κίνδυνος τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται στον τραπεζικό κύκλο, το, ε, κλάδο. Το κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε με συγκεκριμένες τράπεζες και τους λένε ε, στους καταναλωτές Ε, θα προεπιλέξουμε για τον καταναλωτή μία τράπεζα και μετά θα προσφέρουμε εξαιρετικές, ε, εξαιρετικούς όρους. Αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μία ξεκάθαρη δήλωση πως αν αυτή η, αυτό το επόμενο στάδιο συμβεί στην Ευρώπη όπως και στη ΣΥΠΑ, πως εμείς θα το... Ε, θεωρήσουμε παράνομο. Γιατί εμεί τρέχουμε πίσω από τι εξελίξει. Και παρόλο που αυτέ οι εταιρείε καλούνται να ε, πληρώσει ένα υψηλό πρόστιμο, αυτό δεν επιστρέφει την αγορά στην πρωτήτερη της ε, κατάσταση. Νομίζω πως εδώ χτυπάει ε, ένα καμπανάκι και θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και η συνάδελφος. Αν δεν έχουμε άλλες εναλλακτικέ λύσεις, ίσως μια πολιτική δήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλου δεν έχουμε που να ζητούν στη διαδικασία Catch the Eye ε, να ρωτήσουν κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ ε, εκπροσωπείται εδώ από το Γενικό Διευθυντή Ολιβιέ Γκερσά, που πρόσφατα ανέλαβε και ο οποίο ενδεχομένω θέλει να πάρει το λόγο για δύο λεπτά για να απαντήσει. Ξέρω πω τα δύο λεπτά δεν φτάνουν, αλλά σίγουρα θα τα καταφέρετε. Σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συγγήτρια. Είμαι βέβαιο ότι θα με σταματήσετε αν ε, μιλήσω υπερβολικά. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι υπό την αμοιδιότητα που ξαναβρίσκομαι εδώ στην ΕΚΟΝ. Ξέρω ότι πολλοί από εσά έχετε εργαστεί για πολλέ ε, ώρε και ειδικά νύχτα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια νέα θέση, νέα νομική βάση, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε την εξαιρετική συνεργασία και αλληλεπίδραση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και του Κιώδη για την έκθεση. Κάποια σχόλια και καθώ απευθύνομαι σε εσά, κύριε Σιγήτρια, θα συνεχίσω στα γαλλικά. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι προφανώς ε, βασική πολιτική της Ένωσης, επιδιώκει τους στόχου των γενικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσαρμόζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού στις εξελίξεις της οικονομίας και ειδικότερα στις τεχνολογικές εξελίξεις. Το είπαμε παρκώς προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι μεν ε, μια πολιτική μεταξύ άλλων, αλλά οι υποθέσεις ανταγωνισμού ε, έχουν και νομικό χαρακτήρα. Ε, απαιτείται ισότητα στις διαδικασίες όσο και στην εφαρμογή των ουσιοδών κανόνων. Και θέλω να χαιρετήσω λοιπόν θετικά τα όσα υπόθηκαν ε, για να μην είμαστε υπερβολικά παρεμβατικοί ε, σε επιμέρους υποθέσεις. Ε, θα έλεγα στα αγγλικά, αν η πολιτική ανταγωνισμού είναι πραγματική πολιτική, είναι πολιτική, αλλά δεν πρέπει να είναι πολιτικοποιημένη. Είμαστε ευγνώμονε για την υποστήριξη του κοινοβολίου αυτού, ούτω ώστε να παρέχει επαρκή μέσα στην Digicom και με τα πρότυπα, αλλά και σε πόρου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα φαινόμενα που προκαλεί η ψηφιοποίηση. Αντιμετωπίζουμε το θέμα πολύ σοβαρά και προσπαθούμε να βρούμε διδέες αυτή τη στιγμή για να προσαρμόσουμε τους κανόνες μας να δούμε πώς θα τους εφαρμόσουμε, πώς θα προσαρμόσουμε δηλαδή τους κανόνες ανταγωνισμού και τι πρέπει να γίνει και στην τομεακή νομοθεσία. Διότι αν δείτε στο παρελθόν, κάθε φορά που σημειώσαμε επιτυχία ήταν διότι καταφέραμε να έχουμε πολιτικές ανταγωνισμού και τομεακούς κανονισμούς ε, να λειτουργούν παράλληλα. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έγινε αυτό, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των μεταφορών. Ε, Τέλος, επειδή έχω περάσει ήδη τα δυο μου λεπτά, θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο Σβεν Γκίγκολτ. Αν ε, η Ρωσία θα μπορούσε να ε, είναι ανθούσα αυτή τη στιγμή αν ε, το μονοπόλιο λειτουργούσε καλά. Οπότε είναι καλύτερο να κρατήσουμε την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα βοηθάει την καινοτομία. Η ανταγωνιστικότητα ε, προέχει επιλογές στους καταναλωτές και τρίτον διότι αποτελεί ουσιώδη στοιχείο ισότητας εντός της ενιαίας αγοράς. Ας μην είμαστε φυσικά αγαθοί. Θα πρέπει φυσικά ε, ή ισιορροί ανταγωνισμού να βασίζονται σε νόμους, αλλά για να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η πολιτική ανταγωνισμού ε, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση την εμπορική πολιτική για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Κύριε Γενική Διευθυντά. Διπλασιάσατε το χρόνο ομιλία σας. Ίσως. Αυτό να δείξει ότι και τα πρόστιμα θα διπλασιαστούν, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντα όλους σας για αυτή την καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας αυτής ανταλλαγή απόψεων και όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι νέα εδώ, αλλά γεμάτη βούληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτελεί ε, το ρόλο του, δηλαδή να είναι συνομοθέτης υπέρ των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και να έχουμε ε, ανταλλαγές απόψε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως σας είπα, έχουμε 345 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Ε, βέβαια είναι δύσκολο γιατί 6.000 ε, χαρακτήρες δικαιούμαστε να συμπεριλάβουμε στις ε, εκθέσεις αυτές, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τα συμπεριλάβουμε όλα. Θα προσπαθήσω πάντως. Ευχαριστώ πολύ τους και όδες και θα συνεχίσουμε μαζί τη συζήτηση και τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε ευρία βάση για συμφωνία και χαίρομαι. Εξάντε, ναι, με ισορροπία Πολύ σημαντικό αυτό. Να συμπεριλάβουμε επίση και πόσο μεγάλη σημασία έχει να ε, ανδριώνονται οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, να επενθυμίσουμε όμως πόσο μεγάλη σημασία έχει το παιδί εφαρμογή της έκθεσης, που πρέπει να μιλάει για τον ανταγωνισμό. Οι άλλοι τομεί μπορεί να γίνεται κάποια μνήα σε αυτούς, αλλά δεν μπορούν να αποτελήσουν και το κεντρικό σημείο, παρόλο που πολλοί θα θέλανε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα και όχι μόνο για τον ανταγωνισμό. Όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής, η πολιτική ανταγωνισμού είναι μία μόνο πολιτική της Ένωσης. Επίσης, καιρότητα της ενίας αγοράς, να μην υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Εννοείται ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνε. αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να του τηρούμε και εμεί του ίδιου μα του αυτού. Ε, πιστεύω ότι θα βρούμε για τον MSM κάποιο συμβασμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνει αποτελέσματα, εννοείται. Όσο πιο γρήγορα μπορώ θα σα στείλω τι πρώτε συμβαστικέ τροπολογίε που προτείνω και πολύ σύντομα θα συναντηθούμε και πάλι για να συζητήσουμε υπενθυμίζω και το χρονοδιάγραμμα. Η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας ε, θα λάβω χώρα 17 και 18 ε, Φεβρουαρίου και τον Μάρτιο θα ψηφίσουμε, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, φαντάζομαι ξέρετε πότε είναι η Ολομέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ και πάλι και συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι το σημείο 24. οικονομικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση 2019. Εισηγητή είναι ο Μπά Έκχουτ από του πράσινου. Έχετε το λόγο για 6 λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Έκχουτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν τα χρειάζομαι τα έξι λεπτά. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε για την εκθέση αυτή. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση τη δικιά μα επιτροπή στην αρμόδια επί επιτροπή που είναι η Επιτροπή Προπολογισμών. Θα μπορούσε να πείτε μόνο γνωμοδότηση. Ναι, αλλά είναι μια πολύ σημαντική γιατί θα είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με όλες τις αλλαγές και με όλες τις ε, νέες προτάσεις πάνω στις οποίες δουλεύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε τι θα πει το Κοινοβούλιο και τι θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότηση αυτή. Είχαμε δύο συναντήσεις με σκιώδεις εισηγητές και από τότε που συνέταξα το κείμενο αυτό είχαμε και προθεσμία για τροπολογίες την προηγούμενη χρονιά είχαμε μια πρώτη συνάντηση και μια δεύτερη τώρα. Στο μεταξύ συνεδεθήκαμε με τους σκιώδεις εισηγητές, τους οποίους και ευχαριστώ γιατί δούλεψαν σκληρά και ιδιαίτερα επικοδομητικά προκειμένου να καταλήξουμε σε νέα συμβιβαστικές προτάσεις από τις 99, ναι πολλά εννιάρια ξέρω. Οι συμβιβαστικές πιστεύω ότι θα διαρθρωθούν γύρω από την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να καταστεί κλιματική τράπεζα και τι χρειάζεται γι' αυτό. Επικεντρωνόμαστε επίσης στις βασικές τροπολογίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει και η συζήτηση για την χρηματοδότηση που καλύπτεται σε μία από τις συμβαστικές τροπολογίες λαμβάζοντας υπόψη μας την μετάβαση, τη μετάβαση των περιφερειών, για παράδειγμα, ώστε να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περιφέρειες στο σημείο κίνησης για την μετάβαση αυτή. Και επίσης μιλάμε για λογοδοσία, διαφάνεια και φορολογικές πολιτικές και καταπολέμηση της νομοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά λοιπόν είναι κάποια ζητήματα τα οποία καλύπτουμε με τις συμβαστικέ τροπολογίες. Όπως είπα, οι διαπραγματεύσει ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες και μπορώ να πω ότι φαίνεται πως όντω θα καταλήξουμε σε νέα συμβαστικέ τροπολογίες με τις οποίες θα συμφωνήσει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Έτσι θα έχουμε μια γνωμοδότηση που θα την στηρίζουμε ευρέως και που θα σταλεί στην Επιτροπή Προπολογισμών. Πιστεύουμε ότι με εννέα συμβιβαστικέ διευκολύνουμε και την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Γιατί από όλες τις 99 τροπολογίες που υποβλήθηκαν ατομικά, περίπου όλες έχουν καλυφθεί από τις εννέα συμβαστικές. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ και πάλι τους κοιόδης εισηγητές για τη βοήθειά τους και με ενδιαφέρει να ακούσω τώρα τη δικιά τους άποψη, αλλά όχι μόνο αυτών και των υπολείπων συναδέρφων που θέλουν να πάρουν τον λόγο όσον αφορά την ΕΤΕΠ. Ευχαριστούμε. Πολύ αποτελεσματικό ήσασταν και πολύ σύντομα τα είπατε. Μπράβο. Σκιώδης τώρα. Francis Fitzgerald. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάνει πολύ καλές συναντήσεις μεταξύ συγητή και σκιωδών. Συμφωνώ Είμαστε κοντά στο τέλος και προσπάθησα στις τροπολογίες να δώσω κάποιες προτεραιότητες. Καταρχήν υποδομές στην Ευρώπη θα πρέπει να προωθηθούν μέσω της ΕΤΕΠ και στην έκθεσή για το 2019 τονίζει πως οι, οι επενδύσεις στις, υποδομές είναι στο 6,1% του ΑΕΠ της Ευρώπης, το χαμηλότερο την τελευταία 20 ετία με τεράστιες επιπτώσεις για, τα, για τις χώρες μας εάν θέλουμε να δρέψουμε τους καρπούς της ψηφιακής ε, νέας εποχής. Νομίζω ότι η ΕΤΕ μπορεί να μας βοηθήσει πολύ προς αυτό το στόχο. Τροπολογίες υπέρ Τη στήριξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να μειωθεί το κενό το χρηματοδοτικό για τι επιχειρήσει αυτέ και το περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται ε, πολύ σε αυτή την έκθεση και κάποιε αλλαγέ που θα πρέπει να κάνει η ΤΕΠ για να το υποστηρίξει. Αναγνωρίζουμε τι δεσμεύσει που έχω αναλάβει στην Τράπεζα για την χρηματοδότηση δράσεων υπέρ του κλίματος μέχρι το 50% ε, μέχρι το 2025 και επίση. Ε, να ε, συμμορφωθούν όλες οι χρηματοδότητες μέχρι το ε, τέλος του 2020 με τους στόχους του Παρισιού. Δίκαιη μετάβαση. Χρηματοδότηση λοιπόν απαραίτητη για να την πετύχουμε. Νομίζω πως όλα αυτά υπάρχουν στους, στις συμβαστικές τροπολογίες και περιμένω και εγώ με χαρά την περαιτέρω συνεργασία για ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ήταν πολύ επικοδομητικός για τις τροπολογίες από όλα τα κόμματα. Ήταν εξαιρετική η ενέργεια στην, ε, ε, και το κλίμα στις συναντήσεις μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ο συνάδελφος Γιωακίμ Σούστερ δεν μπόρεσε να παραβερθεί και μου ζήτησε να διαβάσω ε, τη δική του, τα δικά του σχόλια. Για τους σοσιαλιστές έχουμε τρία σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής. Καταρχήν, ρόλος του δημοσίου ε, για να επιτύχουμε τους επενδυτικούς στόχους που ανακοίνωσε η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εξασφαλίσει πως οι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη στηρίζουν τις προσπάθειες στο μέρο να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Τονίζουμε τη σημασία που έχει η αιρεσιμότητα στην χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΤΕΠ και η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων. Τέλος, θέλουμε να ενισχυθεί ο λόγος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένα μνημόνιο συνεργασίας ή κατανόησης μεταξύ της ΕΤΕΠ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ενίσχυση του διαλόγου ε, και για να ε, ε, απαντήσουμε σε κάποια θέματα που αναφέρθηκαν στην έκθεση. Είμαστε σίγουροι πως θα συνεργαστούμε και θα στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Renew. Έχουμε κάποιον εδώ από τη Renew για να μιλήσει για το θέμα. Nobody from Renew. Όχι, δεν έχουμε κάποιον από Renew. Okay, now we have uh, uh Jessica Stegroot from ECR. Jessica Stegroot από το ECR. Δεν είναι εδώ. Γκουε, υπάρχει κάποιος από την Γκουε. Όχι. Έχουμε μια ερώτηση κατσιδιάει από την Ενικοκέρη. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχω μόνο κάτι που ήθελα να προσθέσω. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζη Επενδύσεων και από τον ε, πυλώνα 3 ε, του ενίου μηχανισμού σταθερο... Ε, δίκες μετάβασης έτσι να διευκολυνθούν αυτά τα δύο μέσα. Εδώ πρέπει να εστιαστούμε στην λέξη δίκαιος. Just. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να τονίσουμε και σε αυτή την εκθέση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρειάζεται προσαρμοσμένα ε, σε επενδύσεις ανάλογα ε, με τις χώρες ε, και τις ιδιαιτερότητες τους και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Δεν πρέπει να αισθάνεται καμία χώρα ή καμία περιοχή ότι όλη η μετάβαση στην πράσινη οικονομία ε, δεν γίνεται επαρκώς. Οπότε ελπίζω να μπορέσει η συγκεντρία να δεχθεί την τροπολογία μου. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Πάμε πίσω στην εισηγήτρια για τα τελικά σχόλια. Στον εισηγητή, συγγνώμη, για τα τελικά σχόλια. Αν δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Τα όσα είπαν οι συναδέλφοι από το ΕΛΚΑ και τους σοσιαλδημοκράτες ε, υπάρχουν ήδη σε όλες τις συμβιβαστικές που έχουμε συντάξει. Το να τονίσουμε δηλαδή τη σπουδαιότητα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του ρόλου που παίζει στη χρηματοδότηση τη Πράσινη Συμφωνία και στην υποστήριξη ε, των στόχων τη να γίνει κλιματική τράπεζα. Ταυτόχρονα τονίζουμε την ανάγκη για δημόσιε επενδύσει. Ιδιαίτερη προσοχή σε έναν μηχανισμό δίκαιη μετάβαση ε, και αυτό υπάρχει σε μία από τι συμβαστικέ τροπολογίε. Τονίζεται, όπω είπαμε εκεί, το ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ περιοχών και πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτές, το στοιχείο αυτό έχει συμπεριληφθεί. Έγιναν μεγάλες συζητήσεις για το πώς θα βελτιωθεί η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κάτι πολύ σημαντικό, όπως είπε, είπαν οι συναδελφοί σοσιαλδημοκράτες και στις συμβιβαστικές λοιπόν υπάρχει και αυτό το στοιχείο. μία συγκεκριμένη συμβιβαστική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Φιτσέρολτ, είναι σημαντικό και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό υπάρξει σε μια από τις συμβιβαστικές. Οπότε πιστεύω συνολικά ότι όλα τα σημεία που ακούσαμε σήμερα το πρωί συζητήθηκαν και στις συνεδρίασεις των σκιωδών και υπάρχουν τώρα στις συμβαστικές που έχουμε υποβάλει. Με αυτό πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ ομαλή ψηφοφορία με ευρεία πλειοψηφία για αυτή την γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα μπορέσουμε να στείλουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Σα ευχαριστώ ξανά όλου και περιμένουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Για να κλείσουμε αυτό το σημείο, να σα υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ στι 6 Φεβρουαρίου και η Ολομέλεια Μαρτίου. Σας ευχαριστώ. Και πάμε πίσω στην αγαπητό πρόεδρο. Στην ε, κανονική πρόεδρο, συγγνώμη. So we can start, uh, the... Ωραία. Είμαστε στο σημείο 25. Πρόκειται για την Τραπεζική Ένωση της έκθεση 2019. Η συγκητή είναι ο Πέντρο Μάρκε από του Σοσιαλιστές. Έξι λεπτά παρακαλώ για την εισαγωγή σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ελπίζω να μην μου χρειαστεί τόσο πολύ για την αρχική παρουσίαση. Και εδώ είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε για την έκθεση αυτή. Πριν από δέκα χρόνια, όπως ξέρετε, η Ευρώπη αντιμετώπισε μια φοβερή κρίση και συμφωνήσαμε για κάποιες από τις αιτίε της ε, κρίσης. Σίγουρα είπαμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η μεγαλύτερη οικονομική κρίση με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, πολύ περισσότερες από αυτές που θα ανέμενε κανείς. Κάποιες χώρες αντιμετώπισαν επιθέσεις στα κρατικά τους ομόλογα και δυσκολεύτηκε πολύ η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την κατάσταση για μερικά χρόνια. Μέρος της ιστορίας είναι και ο ρόλος των τραπεζών και του τραπεζικού συστήματος και πώς συνεισέφερε στην κρίση. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα δεν λειτουργούσαν καλά και αυτός να είναι ο κύριος λόγος της κρίσης. Άλλοι πάλι λένε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την άλλη αντιμετώπισε την κρίση. Πολλοί ε, επλήγησαν. Η Ευρώπη άργησε πολύ να δώσει απάντηση. Μάθαμε πάντως, πήραμε πολλά μαθήματα από αυτή την κρίση. Ε, μάθαμε ότι ο τρόπος που σχεδιάστηκε το ερώ και λειτουργούσε οδήγησε σε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Μάθαμε επίσης ότι σε περίπτωση ασυμμετρικών σοκ χρειαζόμαστε ε, περισσότερα μέσα. Και επίσης ότι στην νομισματική ένωση έτσι όπω την έχουμε υπάρχει αλληλεξάρτηση στο οικονομικό σύστημα με αποτέλεσμα να είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε μια τραπεζική ένωση που να λειτουργεί ικανοποιητικά. Μάθαμε επίσης ότι οι τράπεζες ε, μπορεί και να πτωχεύσουν. Και όταν είναι μεγάλες αυτές, ήταν οι φορολογούμενοι αυτοί που έπρεπε να πληρώσουν την ύφη. Δεν θέλουμε όμως αυτό να ξανασυμβεί. Με αυτό και άλλα μαθήματα που πήραμε από την κρίση ξεκίνησαν οι μεταρρυθμίσεις. Όμως μετά συνεχίσαμε η κρίση λίγο πολύ λίγο σταμάτησε, άρχισε κάποια ανάπτυξη στην οικονομία. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάποια στιγμή θα ξανά έχουμε κρίση. Και αν δεν ολοκληρώσουμε τώρα τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Τα ζητήματα βέβαια οδηγούν μερικές φορές σε διαφωνίες, ε, κάτι το οποίο μας εμποδίζει να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις. Οπότε δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Στόχος της έκθεσης αυτής λοιπόν είναι για διάφορα ζητήματα να ε, προχωρήσει Δίνοντα τη δυνατότητα για συνένεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμού και έτσι να φανεί η σαφή βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσει αυτές. Τα πράγματα δεν πρόκειται να λυθούν από μόνα τους αν απλώς δεν τα συζητάμε. Όχι, η Τραπεζική Ένωση ξέρουμε ότι δεν έχει τον τρίτο της πυλώνα που είναι το EDIS, το σύστημα δηλαδή εγγύσεων καταθέσεων και χρειαζόμαστε επίσης περισσότερα και από το ε, Ταμείο Το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν υπάρχει τίποτα προσυζήτηση πια. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήσαμε, που ακούστηκαν σε διάφορες ακρόσεις ε, που είχαμε με χρηματοπιστωτικά δρήματα πριν από την πρώτη παρουσίαση της έκθεσης. Και θα λαμβάνουμε υπόψη μα οι συνάδελφοι σιώδη, οι συγητέ ε, και εγώ στι προτάσει μα. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ευχαριστώ για τι τροπολογίε που υπέβαλαν οι Σκιώδη αλλά και άλλοι συνάδελφοί μα. Θα τι λάβω υπόψη μου, όπω γνωρίζετε. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση σκιωδών που ήταν επικοδομητική και είμαι σίγουρος ότι και η δεύτερη θα είναι επικοδομητική και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβασμού. Σας ευχαριστώ όλους, για άλλη μια φορά τους σκιώδεις, τους συνεργάτες, τη γραμματεία για την ε, στήριξή τους μέχρι τώρα και είμαι σίγουρη ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας να επιτελέσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή σας αυτή. Πηγαίνουμε στους σκιώδεις, πράγματι. Ελκ, η Ντανούτα Χούμπνερ. Έξι λεπτά έχω κι εγώ. Τρία, τρία, τρία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον Πέντρο Μάρκε. Και όχι, δεν το λέω αυτό απλώ επειδή πάντα λέμε ευχαριστώ στου συναδέλφου, αλλά γιατί πιστεύω ότι είχε αυτή την εξαιρετική ιδέα να οργανώσει με την γραμματεία, του οποίου επίση ευχαριστούμε, διάφορε ακροάσει όπου προσκαλέθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή ε, άλλους που έχουν να κάνουν με αυτά τα θέματα και έτσι ακούσαμε τη δικιά του αξιολόγηση. Ήταν πολύ χρήσιμο. Και είναι καλό επίση να το έχουμε υπόψη μα και για το μέλλον και για άλλε εκθέσεις να ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Ευχαριστώ επίσης όλους του συνεδέρφου, όχι μόνο τους Κιώδης, αλλά και άλλους που με τις τροπολογίες τους συνεισέφεραν σημαντικά στις συζητήσεις και στην διεύρυνση των ε, απόψεών μας. Πράγματι, η έκθεση αυτή, όπω είπε και ο Πέντρο, ακολουθεί το ίδιο μοντέλο με τις προηγούμενες, δηλαδή παρακολουθεί λίγο την ιστορία, την εξέλιξη της Τραπεζικής Ένωσης. Κάτι το οποίο μας βοηθάει να εντοπίσουμε τις προσκλήσεις που μένουν, τις δυσκολίες, τις αδυναμίες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον τρίτο πυλώνα αλλά και με άλλα θέματα σημαντικά. Πάντως, οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση πέρασαν την δοκιμασία γιατί τα κατάφεραν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά σίγουρα πρέπει να στραφούμε προς το μέλλον και να φροντίσουμε να είμαστε ανθεκτικοί εν ώψη μιας επόμενης ενδεχομένω κρίσης. Τώρα για διάφορα ζητήματα νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε λίγο πολύ σε μια κοινή προσέγγιση, σε ένα συμβασμό θα συνεχίσουμε με το ίδιο αυτό πνεύμα. Νομίζω ότι συμφωνούμε για το πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την προστασία των ε, καταναλωτών σε περίπτωση που κάποια ε, τράπεζα πτωχεύσει, να νιώθουν ότι οι καταθέσεις τους είναι εγγυμένες, και επίσης είναι κοινή και η ανησυχία για το θέμα της κερδοφορίας και τον ανταγωνισμό του ευρωπαϊκού οικονομικού τομέα των τραπεζών. Κοιτούμε λοιπόν και το θέμα των χαμηλών επιτοκίων, του σημερινού περιβάλλοντος, της τρέχουσας κατάστασης, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κλπ. Επίσης, εξετάζουμε και το δίλημα για τον επιμερισμό κινδύνου ή το μηδενικό κίνδυνο. Προσπαθούμε να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο. Αυτό όμως που παραμένει ως θέμα είναι μια καλά σταθμισμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη δυνατότητα της Ένωσης να συνεισφέρει σε ασύμετρα σοκ σε περίπτωση κρίσεων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρω αν θα βρούμε μια κοινή λύση. Αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί σε αυτή την έκθεση. Υπάρχουν και πολλά άλλα που εξετάζουμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε έγκαιρα. Να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Με επιτυχία. Ώστε να ψηφίσουμε καλά στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τρία λεπτά, Renew, Σκιώδης. Εγώ απλώς θα επαναλάβω τις ευχαριστίες μου ε, για τον τρόπο με τον οποίο ανέλαβε αυτό το καθήκον και για το προσωπικό που τον βοηθάει, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε όταν μιλάμε για Τραπεζική Ένωση είναι τεράστιε. Γιατί αν μιλά κανεί αφηρημένα, όλα μπορούν να λυθούν. Όταν μιλά για την πολιτική διάσταση πίσω από του ορισμού και τα συμφέροντα των κρατών μελών, τότε όλα περιπλέκονται. Και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα τα όσα προτείνεται για την ακαιρεότητα του τραπεζικού συστήματο που στηρίζεται από υποπτία, από ε, προληπτική δράση, από ε, διατάξει και και να μην ξεχνάμε πως πρέπει να υπάρχει κεφάλαιο, το οποίο, να υπάρχουν κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα για την πραγματική οικονομία με λογικά επιτόκια, με προστασία και των καταναλωτών αλλά και των φορολογουμένων σε περίπτωση που η κατάσταση ε, χειροτερεύσει και να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε με τις πολιτικές που θα, εφαρμόσει το, θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Αν αμφίβολα δεν υπάρχει αυτή η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρώπη και από τη στιγμή της κρίσης οι τράπεζες απλώς ε, κλείστηκαν στα εθνικά του σύνορα και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την τραπεζική δραστηριότητα μέσα στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε εθνική εποπτεία και όχι ευρωπαϊκή εποπτεία. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμεθα από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών για να ε, φέρουν σε πέρα στην εποπτεία του τραπεζικού του συστήματο. Και έχουμε ε, και εποπτεία και εξυγίανση, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν κυρίως μέσα στα κράτη-μέλη, το οποίο σημαίνει ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη που αισθάνονται στον εαυτό τους οι τράπεζες για να ξεφύγουν από τα εθνικά σύνορα και να δράσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα μεγάλα θέματα είναι η προστασία των φορολογουμένων και το ε, θέμα ε, εδώ είναι τι γίνεται με ε, ε, τις τράπεζες ε, και τα κρατικά ομόλογα που είναι αλληλένδετα ε, σε εποχές κρίσης και αλληλοεξαρτώμενα. Αυτό έχει να κάνει με τα διάφορα κόμματα και τα κράτη-μέλη και τις κυβερνήσεις τους, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πριν μπούμε στη συζήτηση ε, της βελτίωσης τραπεζικής αγοράς. Δηλαδή, μια, οποιαδήποτε κατάρρευση σε ένα κράτος μέλος, είτε ε, στα κρατικά ομόλογα, είτε στις τράπεζες, οδηγεί σε συνολική κατάρρευση αυτή τη στιγμή. Επίσης, για την εποπτεία, το ξέπλυμα χρήματος είναι ζήτημα είναι ζήτημα ηθικό και για τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν πως έχουν ένα στεναρό όργανο έρευνας κατά του ξεπλήματος γιατί οι οδηγίες προέρχονται από την Ευρώπη, αλλά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες και εκεί θα πρέπει τα συστήματα να είναι ισχυρά και να βελτιωθούν. Δεν μπορεί εμείς να πιστεύουμε πως η κατανομή κινδύνου θα γίνει ο κανόνας αν τα κράτη-μέλη και οι φορολογούμενοι στην Ευρώπη κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα όταν μια τράπεζα α, ε, ε, καταραίει ε, επειδή οι διατάξεις για να εξασφαλιστούν οι τράπεζες από το ξέπλυμα χρήματος δεν έχουν εφαρμοστεί. Μείωση επίσης των επισφαλιών και εκεί πολύς χρόνος μένει μέχρι να λύσουμε το θέμα της κατανομής κινδύνου Πιστεύω πάντως που αν συνεχίσουμε το διάλογο και τη συζήτηση θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδους συνένεση. Αλλά χρειάζεται να έχει λεπτομέρειες αυτή η συνένεση για να επιβάλλουμε στα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσουν στις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank uh, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κελνέρ για τους ε, πρασίνους. Ο κ. Σορτασούν, ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση και τον ε, εισηγητή που καταφέρει να επιτύχει ευρεία πλειοψηφία στις συναντήσεις ε, σκιωδών. Υπάρχουν κάποιες κάποια στοιχεία στι τροπολογίες μου. Μετά από την οικονομική κρίση εξακολουθούμε να βλέπουμε πολλά στους χρηματοοικονομικούς μα κανονισμού που δεν προλαμβάνουν την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εμεί έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίες που ασχολούνται με αυτέ τι προκλήσεις που απομένουν όχι μόνο την ύπαρξη των ιδρυμάτων του Big to Fail που παραμένουν βασικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Τα πρόσφατα χρόνια έχουμε προχωρήσει πολύ στη μέση του κινδύνου στο οικονομικό μα σύστημα το νέο πλαίσιο ανάκτησης και εξυγένσης ε, είναι κάτι πολύ καλό, αλλά είναι αργή η πορεία προς το καταμερισμό κινδύνων. Είναι σημαντικό λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία για να υπάρχει μια ισχυρή, σταθερή τραπεζική ένωση, οπότε χρειάζεται να το πούμε ε, ρητά, ειδικότερα σε αυτή τη στιγμή της συζήτησης, κάτι απολύτως αναγκαίο στην έκθεση. Σήμερα ψηφίσαμε τους νέους διορισμούς για την ΕΑΤ, και τους άλλους οργανισμούς. Οπότε εδώ στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρουμε την έλλειψη ε, ισότητας του φύλου. Μετά από όλες τις υποσχέσεις ε, που είχαμε από την Κομισιόν πρέπει να γίνουν επιτέλους οι μεταρρυθμίσεις ώστε να είναι η τελευταία φορά αυτή που ε, διορίζονται μόνο άντρε. Χρειάζεται να έχουμε μια σαφή αναφορά σε αυτό ότι δεν μπορούμε πια να δεχτούμε short list που να περιλαμβάνουν μόνο άντρες για τους οργανισμούς μας. Επίσης, εμείς θέλουμε να τονίσουμε τις βιώσιμες, τα βιώσιμα οικονομικά, την ταξινομία. Συζητήσαμε σήμερα και την ψηφίσαμε και αυτό ήταν σημαντικό βήμα. Απευθύνουμε και έκκληση για μια βασική ταξινομία που είναι απαραίτητη. Μια προτεραιότητα τη ομάδα μα είναι να διασφαλίσουμε επίση την προστασία των καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του και οδησυγητέ και τον, και τον εισηγητή που δέχθηκαν να το συμπεριλάβουν ε, αυτό στην έκθεση τη τροπολογη 31 31-32-165 αναφερόμαστε στη σκανδαλώδη συμπεριφορά των τραπεζών προ του καταναλωτέ ε, και προτείνουμε εναλλακτικέ. Επίση θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προστατευτούν ε, οι ευάλωτοι δανειολήπτε στεγαστικών δανείων οπότε θέλουμε να δοθεί ε, κάποια εγγύηση για την προστασία των δανειοληπτών. Σύμφωνα και με τις συζητήσεις που κάνουμε για τους διαφορούς κανονισμούς σήμερα είναι σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη δράση για το ξεπλήμα μαύρου χρήματο. Και τέλος, στην τροπολογία 172 θέλουμε καλύτερη ρύθμιση των κινδύνων της κοιόδου τραπεζικού συστήματος για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένες αυτές οι δραστηριότητες σε μεγάλου κινδύνους με χαμηλά στάνταρ και θέλουμε να ρυθμιστεί επιτέλους αυτός ο τομέας. Συνολικά θα έλεγα ότι όλες αυτές οι ιδέες θα τροφοδοτήσουν συζητήσεις ε, και σκέψεις ε, για κάτι που ήδη θεωρούμε εξαιρετική βάση για τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας για το ID. Ευρωζοβάρνα, αλλά δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει για το ID. Όχι. Οπότε, από το ECR, που είναι σκιώδης. Κάποιος που θα θέλει να μιλήσει για το ECR. Όχι. Μάρτιν Σιντεβέλ από την ΚΟΕ. Είναι εδώ, τον βλέπω. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι επικοδομητικός ο τρόπος ε, που εργάστηκε μέχρι στιγμής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι για να υπάρχει μεγάλη συμφωνία σε πολλά θέματα. Εμείς ως Γκουε περιοριστήκαμε σε πολύ συγκεκριμένες ε, τροπολογίες στη διαδικασία μέχρι τώρα, ώστε να ενισχύσουμε ε, κάποια σημεία της έκθεσης. Πρώτον, κατά την άποψή μας στον τραπεζικό τομέα, από τότε που ξεκίνησε η ε, κρίση δεν αντιμετωπίσαμε επαρκώς τα δομικά προβλήματα στο παρελθόν. Ε, υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις, ε, κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σε περίπτωση νέας κρίσης ε, θεωρώ ότι οι μηχανισμοί εξυγίανσης είναι ανεπαρκείς, αδύναμοι. Δηλαδή σε περίπτωση νέας χώρας πάλι θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Για μας είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα του too big to fail, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν οι πρώτε πρώτες προσεγγίσεις εδώ στην έκθεση και χαιρόμαστε για αυτό, αλλά θέλουμε να ενισχυθούν κι άλλο. Και δεύτερο, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, καθώς ε, περιορίζεται ο τομέας, ε, θα πρέπει τα δημόσια και περιφερειακά ιδρύματα στον τραπεζικό τομέα να παίζουν ε, βασικό ρόλο. Έτσι πρέπει ε, κάποια από τα σχέδια της Κομισιόν δηλαδή για την ε, συνέχιση της παγίωσης του τραπεζικού τομέα θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη. Οι τεράστιες ε, συγχωνεύσεις για παράδειγμα θα πρέπει να, που, θέλει να διευκολυνθούν και για την ασφάλεια των καταθέσεων αν αυτή σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της παγίωσης ε, και της καταμερισμού κινδύνου ε, και ε, στις τράπεζες και στους κεφαλαγορές. θα πρέπει να ακολουθούν και τα περιφερειακά και τοπικά ιδρύματα επίσης και εμείς θα κάνουμε προτάσεις για το πώς αυτό θα οργανωθεί στο μέλλον. Αλλά πιστεύω ότι από αυτά που άκουσα μέχρι σήμερα ότι έχουμε καλές συμβιβαστικές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για μας. Ε, υπάρχουν δύο σημεία που για μας είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα διαπραγματευτούμε περισσότερο. Πρώτον, ε, περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα είναι λάθος, είναι κόκκινη γραμμή. Ε, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε λοιπόν. Ε, μπορεί και η ψήφο μα υπέρ τη έκθεση να εξαρτηθεί από αυτό. Και μετά, όταν μιλάμε για περισσότερη μείωση των κινδύνων, ε, μιλάμε βέβαια πολύ σωστά να μειώσουμε του κινδύνου ε, των κρατικών ομολόγων. Ε, να τα ενισχύσουμε όλα αυτά μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα. Αλλά πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και αναμένω επικοδομητικές συζητήσεις και με τον εισηγητή και με τους λοιπούς και Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Μάρτιν. Δεν βλέπω κανένα για το Κατζέι. Οπότε, κύριε Μάρκες, θέλετε να καταλήξετε σε συμπεράσματα μετά από τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ. Τίποτα, μεταπλώσω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδει συζητητέ, όλους όσοι πήραν το λόγο και η επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη εβδομάδα, θα είναι σκιωδών και εκεί πιστεύω ότι θα πλησιάσουμε περισσότερο στους συμβιβασμούς και ελπίζω ότι στο τέλος να υπάρξει μια ε, συμφωνία πάνω σε αυτούς τους συμβασμούς για την προστασία των καταναλωτών και των φορολογούμενων για να αποφύγουμε την επόμενη συστημική κρίση και να διαθέτουμε τα εργαλεία προς αυτό το σκοπό για να μην ε, υποστούμε συνέπειες στην ε, Ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, τελικά πρόκειται για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η θέση του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι ισχυρή ώστε οι άλλοι θεσμοί, το Συμβούλιο, όλους ιδιαίτερως να καταλάβει ότι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχουν τίποτα άλλο πέρα από την προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Πρόκειται για την προστασία των πολιτών μας. Και δεν θα σταματήσουμε παρά μόνο αν, πετύχουμε, αν το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μάρκε. Ξέρω ότι υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και ενότητας μεταξύ των εισηγητών. Αυτό είναι καλό νέο κάπου 300 τροπολογίες έχουν υποβληθεί. 17 και 18 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Έτσι ολοκληρώνεται και το σημείο 25, σημείο 26, διάφορα, δεν υπάρχουν διάφορα και τέλος η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις 27 Ιανουαρίου, Δευτέρα. Οπότε θα τα πούμε τότε, εκείνη τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιστροφή στις χώρες σας και καλό Σαββατοκύριακο.